τοποθέτηση με τις απαντήσεις. Επτά είναι οι προτάσεις ψηφίσματος. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Ψηφίζουμε την Πέμπτη τα ψηφίσματα αυτά και θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τεχνικού